περνάμε στην δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν για τις σχέσεις με την Ελβετία. Υπενθυμίζω πως μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων δεν θα έχουμε εδώ πέρα την διαδικασία και HDI ούτε μπλε κάρτες. Για το Συμβούλιο ο κύριος Κούρκουλας έχει το λόγο. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίου στην Ελβετία στι 9 ε, Φεβρουαρίου, όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία για την μετανάστευση, δημιούργησε και διαμόρφωσε μια καινούργια κατάσταση. Αντόπιν αυτών των τριών δημοψηφισμάτων που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια στην χώρα, ο λαό έχει εγκρίνει την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τα κρατημέλη. Οπότε το αποτέλεσμα αυτού του δημοσιοφίσματο δεν ήταν ε, κάτι το ευνοϊκό, κάτι θετικό για την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Οπότε, εν προκειμένου, αποφάσισαν με κάποια οριακή πλειοψηφία οι Ελβετοί να αλλάξουν το σύνταγμα του. Και έτσι, μέσα σε τρία χρόνια από το δημοψήφισμα να θεσπίσουν κάποιε ποσοστώσει για του αλλοδαπού, για τι ε, άδειε παραμονή και άδειε ασκήσεω επαγγελματο. Και μετά την ε, αναθεώρηση αυτή του ε, δημοψηφίσματος, ε, η, η, τα ελευθερία επαγγέλματα, οι υπάλληλοι και οι οικογένειές τους πρόκειται να φύγουν από αυτά τα μέτρα. Επίσης, το νέο άρθρο του συντάγματος απαγορεύει την σύναψη νέων συμφωνιών και επίσης υποχρεώνει την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί εκ νέου κάποιες διεθνείς σύμφωνες οι οποίες πρόκειται να αντιβαίνουν ή στις νέες διατάξεις του συντάγματος οι οποίες κατάφορα αντιτίθενται στην Συμφωνία ΕΕ Ελβετίας του 2002 όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Για να υπάρξει συμμόρφωση με το νέο άρθρο του συντάγματος, η Ελβετία θα πρέπει να ζητήσει να γίνει εκ νέου διαπραγμάτευση της σχετικής συμφωνίας, τόσο ώστε να είναι δυνατόν να ε, θεσπιστούν αυτές οι ποσοστώσεις για μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες που στηρίζουν την ε, ενιαία εσωτερική αγορά. Είναι αδιαχώριστη και αδιαίρετη αυτοί οι τέσσερις πυλώνες. Η χώρα, η Ελβετία, τα τελευταία 20 χρόνια έχει συμμετάσχει σε όλο ένα και περισσότερες τομείς της εσωτερικής αγοράς. Επίσης έχει διατυπωθεί η θέληση να ε, ανοίξουν διαπραγματεύσεις και για άλλους τομείς. Οπότε, κατόπιν των όσων έγιναν τώρα δεν είναι δυνατόν να προσδοκάει η Ελβετία ε, εμείς να επικυρώσουμε ε, αυτή την απόφαση όσον αφορά την διακίνηση των προσώπων. Έχουμε όμως και άλλες περιπλογές. Η δεύτερη διακίνηση των προσώπων και σχετική συμφωνία συνδέεται με κάποια ε, ρήτρα γκυλοτίνα με έξι άλλες συμφωνίες που έχουμε αυτή τη χώρα που καλύπτουν μεταξύ άλλων μεταφορά διαξηράς, θαλάσσης, ε, ε, μεταφορά εμπορευμάτων, ε, τις δημόσιες συμβάσεις προμηθείας, οπότε εάν έχουμε κάποιο είδους λήξη αυτών των, των συμφωνιών, θα έχουμε λήξη όλου του πακέτου, το οποίο θα καταπέσει. Οπότε το θέμα είναι το πώς θα προσχωρήσει τώρα η χώρα ή στο κεκτημένο τη δεύτερη σύμβαση του Δουβλίνου. Μα και αυτό θα πρέπει τώρα να θεωρηθεί αν έχουμε τέτοιο περιορισμό τη ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με το ότι το πρωτόκολλο το οποίο ε, παρεκτείνει την ε, ισχύ αυτού του, του, πρωτοκόλλου για τα πρόσωπα στην Κροατία δεν έχει ε, υποβληθεί Οπότε δεν έχει υπογραφεί, συγγνώμη. Οπότε το θέμα είναι πώ εν του δημοψηφίσματο θα μπορέσει να προσυπογράψει η Ελβετία αυτή την, την συμφωνία που αφορά την Κροατία. Δεν μα έχει ακόμα κοινοποιήσει κάτι σχετικά η κυβέρνηση τη χώρα, αλλά υπάρχουν ενδείξει ότι κατά το μάλλον ήταν δεν θα γίνει αυτή η υπογραφεί. Οπότε θα πρέπει να αποφευθούν οι δυσμενείς διακρίσεις. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη διαμόρφωση μιας τέτοιας κατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνδέσει την συμμετοχή της Ελβετίας στο Έρασμο ε, ΣΥΝ και ορίζον 2020 με την συμμετοχή της Κροατίας όσον αφορά τη συμφωνή την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Οπότε, με αυτό το δημοψήφισμα και αφού ακόμα δεν έχουμε λάβει κάποιο είδου κοινοποίηση για την προσυμπογραφεί αυτό το πρωτοκόλλο, εμείς ως ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ακυρώσει τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων. Οπότε, από το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει τις σχέσεις με τη χώρα να τις βάλει σε μια νέα βάση. Θεωρούμε ότι αυτό το περίπλοκο σύστημα των 120 τομιακών συμφωνίων με την χώρα έφτασε τα όρια του. Οπότε θα πρέπει αυτό το σύστημα, αυτό το σύνολο να πλαισιωθεί από ένα ε, θεσμικό ε, ε, θεσμικό καινούριο πλαίσιο. Οπότε τον Μάη του 2012 είχε ζητηθεί να δούμε πώς θα περιληφθεί κάποια πρόοδος και πώς θα προχωρήσουν κάποια εκκρεμή θεσμικά ζητήματα. Κατόπιν μια σειρά ε, συνομιλιών ε, επεξηγηματικών, τον Νοέμβριο του 2013 η Κομισιόν υπέβαλε στο Συμβούλιο μια διαμοτευτική εντολή όσον αφορά αυτό το θεσμικό ε, πλαίσιο για τι σχέσει με την Ελβετία. Και σε τεχνικό επίπεδο υπετέχθη συμφωνία. Το Συμβούλιο τώρα σκέπτεται το πώς θα μπορέσει να προωθηθεί αυτή η εντολή διαμοντευτική κατόπιν του δημοψηφίσματος. Πρόκειται να παρακολουθήσουμε προσεκτικά τις εξελίξεις στη Σουηδία κατόπιν της υλοποίησης του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Έχει πει η Ελβετία ότι πρόκειται να υποβάλει ένα ε, πρόγραμμα ε, υλοποιήσει μέχρι τον Ιούνιο. Και επίση θα νομοθετήσει μέχρι το τέλο του εναστότο έτου. Αλλά θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το ελβετικό πρόγραμμα υλοποίηση του δημοψηφίσματο και να προβληματιστούμε για τα περαιτέρω διαβήματα στα οποία θα προβούμε από πλευρά μα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, εν κατακλείδη θα πρέπει να σα πω ε, ότι ενώ σεβόμεθα την απόφαση του ελβετικού λαού, οι σχέσει μα με την Ελβετία τώρα ε, έχουν μπει σε δοκιμασία λόγω του αποτελέσματο αυτού του δημοψηφίσματος τη 9 η Φεβρουαρίου. βεβαιω χαιρετίζουμε το γεγονο ότι η Ελβετία επιβεβαίωσε μετά τον ψηφισμό ότι πρόκειται να τηρήσει τις διεθνείς τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τις τη συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω συνεχίζει να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις ε, μακραίωνε σχέσεις με την Ελβετία και είμαι θα έτοιμοι να αναζητήσουμε λύσεις στην παρούσα δύσκολη κατάσταση. Αυτό θα απαιτήσει χρόνο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να σεβαστούμε τις ε, ιδέες, τις αρχές μας και δεν θα πρέπει να έχουμε μια περιπτωσιολογική προσέγγιση στην ευρωπαϊκή ε, ολοκλήρωση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό κατά παραγγελία και θα πρέπει οπωσδήποτε να μείνει προσλωμένοι στις βασικές θεμελιώδες μας αξίες. Σας ευχαριστώ, ο πρώτος ο κύριος Σάντορ. Και εγώ θα ήθελα να πω λίγα λόγια ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις μετά το δημοψήφισμα στην Ελβετία στις 9 Φεβρουαρίου. Η Συμφωνία Ελεύθερης Κυκλοφορίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας επιτρέπει στους πολίτες μας να παραμείνουν στην Ελβετία και να εργαστούν στην Ελβετία ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι. Υπάρχουν 450.000 ε, Ελβετοί πολίτες που μπορούν να διαμείνουν στην Ευρώπη και 1.200.000 αντίστοιχοι ε, Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν στην Ελβετία. Και σε καθημερινή βάση υπάρχουν 350.000 ε, μετακινούμενοι για να εργαστούν στην Ελβετία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις ε, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις ε, μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά και προβαίνουμε όλοι σε εμπορικές ε, συναλλαγές. Αυτά βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην αμοιβαιότητα. Όμως το δημοψήφισμα της 9ης Φεβρουαρίου αμφισβητεί την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Ε, ανέφεραν στην Επιτροπή ότι χρειάζονται χρόνο για να δουν τις περαιτέρω εξελίξεις. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο διαθέτει τρία χρόνια για να εφαρμόσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής. Ε, στο μεταξύ και οι δύο πλευρές θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρούν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της ε, παρούσας συμφωνίας. Πάκτα σουν σερβάντα. Η συμφωνία είναι συμφωνία και δεν μπορούμε να έχουμε επιλεκτική εφαρμογή της συμφωνίας. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να ακούσει τις προτάσεις Ελβετίας τις οποίες δεν έχουμε δει ακόμα ε, επιτάπητος. Το μπαλάκι είναι στο δικό τους γήπεδο. Πιστεύουμε όμως ότι αυτή η βασική η θεμελιώδης αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεών μας. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς ε, η μεταναστευτική πολιτική θα ήταν συμβατή με την συμφωνία αυτή για την πλήρη ε, ελεύθερη διακίνηση των πολιτών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας. Δεν μπορούν να υπάρχουν ποσοστώσεις σε αυτές τις μετακινήσεις, διότι η αρχή αυτή δεν μπορεί να αποδεσμευθεί από τις άλλες αρχές. Πρόκειται για πακέτο συμφωνιών το οποίο θα πρέπει να ε, τηρηθεί. Δεν μπορεί να υπάρχει επιλεξιμότητα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συνέπειες επί του συντάγματος της Ελβετίας ε, μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θα εξετάσει κατά πόσο μπορεί να διαπραγματευτεί ένα αρχικό πρωτόκολλο το οποίο θα διευρύνει και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών με την Κροατία. Η Κροατία είναι σαφής ότι περιμένει αυτή την ε, επέκταση Τη της συμφωνίας και δεν μπορεί να δεχτεί την ε, επιλεκτική μεταχείριση των απορριτών. Πιστεύουμε ότι μέχρι τις αρχές Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το πρωτόκολλο. Για να αποφύγουμε τέτοιες διακρίσεις, το Συμβούλιο ε, έλαβε υπόψη και την ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελβετίας στον ορίζοντα 2020 και το Erasmus που συνδέονται άμεσα με το πρωτόκολλο αυτό. Άρα οι διαπραγματεύσεις δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι ότου ε, συναυθεί αυτό το πρωτόκολλο και ολοκληρωθεί από την Ελβετία επί χάρτου. Ελήψη Διεθνούς Συμφωνίας για να ορίσουμε την ε, σύνδεση της Ελβετίας στον ορίζοντα 2020. Η Ελβετία δεν συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα ως συνεργαζόμενη αυτό σημαίνει ότι η ενδεχόμενη συμμετοχή των ελβετικών ε, αρχών ε, το 2014 στον ε, ορίζοντα 2020 εξαρτάται. Θα πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα της, του δημοψηφίσματος. Δεν μπορούμε πλέον να δεχτούμε την ευρωπαϊκή δικτατορία της Ευρώπης. Ζήτω η Ομοσπονδία, ελευθερία των λαών. Τέλος τη δικτατορία της Ευρώπης. Κύριε Μποργκέιτσιο, αποβάλλεστε από την αίθουσα. Κύριε Μποργέτσιο, παρακαλώ να φύγετε από την αίθουσα τη Ολομέλεια. Uh, Κύριε Μποργέτσιο, παρακαλώ εγκαταλείψτε την αίθουσα. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ συνεχίστε. Ε, αναφέρθηκα στο πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης. Ε, η Ελβετία είναι εκπρόθεσμη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα το 2014. Αυτό σημαίνει ότι το 2014 η Ελβετία δεν θα συμμετάσχει στο Erasmus Plus ε, ισότιμα με τα άλλα κράτη-μέλη και η συμμετοχή της θα περιοριστεί σε διαδικασία συνεργασίας όπως ισχύει για οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Αυτό δεν αποτελεί τιμωρία ή κύρωση για την απόφαση του εκλογικού σώματος, αλλά για την επιλογή που έκανε η ίδια η Ελβετία, η οποία ήταν γνωστή εκ των προτέρων. Δεν μας εκπλήσει βεβαίως και κανένας δεν θα ήθελε να διακόψει το διάλογο, ο οποίος θα συνεχιστεί επικοδομητικά, ελπίζοντας να εξευρεθεί μια λύση τάχιστα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες και τη μη ολοκλήρωση του Κροατικού ε, πρωτοκόλλου. Εδώ δεν πρόκειται για επιλογή. Επίσης θα πρέπει να είμαι απόλυτα σαφής, κανένας από την πλευρά μας δεν θέλει να λήξει η διαδικασία ελεύθερης κυκλοφορίας και ελευθεριών των πολιτών με βάση το πακέτο που συνήφθη το 1999 δεν θέλουν ε, κάτι τέτοιο οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Ελβετία θα καταβάλει σοβαλές προσπάθειες για να διευρύνει αυτό τον ε, κύκλο και σε ένα χρόνο να μπορέσουμε να πούμε ότι η σχέση με ε, την Ελβετία ήταν στενές και φιλικές όπως πριν από το δημοψήφισμα. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ακολουθούν οι εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Μαγκίνε για 3,5 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Δεν αμφισβητούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ελβετία, ούτε και το δικαίωμα της Ελβετίας ως ε, κυρίαρχης χώρα να αποφασίζει για τέτοια θέματα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αναλύουμε τις συνέπειες σήμερα τη απόφαση αυτή. Η απόφαση ήταν σαφής αν και με μικρή διαφορά 50,3% ήταν υπέρ του δημοψηφίσματος. Και από ό,τι κατάλαβα η στήριξη ήταν πολύ υψηλότερη σε περιοχές όπου, υπήρχαν, ε, ελάχιστη, όπου υπήρχε ελάχιστη κινητικότητα Ευρωπαίων πολιτών. Βεβαίως ε, πρόκειται για μια συμφωνία η οποία ανάγεται στη δεκαετία του 1970 και άλλες συμφωνίες του 1999 και 2004 επίσης ε, και η συμφωνία του 2002 η οποία συμπεριλάμβανε την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, τα δικαιώματα σημαίνουν και υποχρεώσεις. Και ήταν σαφές ότι ε, περιμέναμε και εμείς από τους Ελβετούς όταν ε, υπογράφουμε αυτές τις συμφωνίες. Μπορεί κανείς να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ως μια επιθυμία να τερματιστούν οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι σαφές πως αυτό δεν συμβαίνει, γιατί ψήφισαν για ένα και ένα μόνο στοιχείο της σχέσης τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να περιορίσουν την πρόσβαση στην Ελβετία για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η ελεύθερη διακίνηση είναι θεμελιώδες τμήμα των συμφωνιών μας με την Ελβετία και θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν έχει δηλώσει και πάρα πολλοί επίτροποι σήμερα το πρωί πως είναι αδύνατον να περιοριστεί η ελεύθερη μετακίνηση και να περιμένουν ότι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν την ελεύθερη διακίνηση ε, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου αντιλαμβάνονται πλέον, ε, αντιλαμβάνεται η ελβετική κυβέρνηση πως υπάρχει μια συστημική αλλαγή από το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος. Και αντιλαμβάνομαι πως λόγω της αβεβαιότητας κάποιες επιχειρήσεις αναζητούν ε, πιθανή μετακίνηση εκτός Ελβετίας λόγω της αβεβαιότητας αυτής. Οι Ελβετοί εταίροι μας θα ήθελαν να διαλέγουν σε ποιον επιτρέπουν πρόσβαση στο πλαίσιο της ελεύθερης μετακίνησης και ακούγονται και ποσοστώσεις. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Οι ποσοστό είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο συμφωνήσαμε με τους Ελβετού. Υπάρχουν τρία χρόνια περιθώριο μέχρι να εφαρμοστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αλλά ήδη η κυβέρνηση αντέδρασε με το να μην υπογράψει το πρωτόκολλο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επεκτείνει την ελεύθερη μετακίνηση και στους ε, κροάτε υπηκόου. Οπότε απαιτείται και εμείς να πούμε πώς θα ακυρώσουμε τις συνομιλίες για το Εράσμους και τα επιστημονικά προγράμματα και νομίζω πως και οι ευρωβουλευτές από την Κροατία θα ήθελαν να υπρασπιστούμε τα δικαιώματά τους. Τώρα εγώ δεν πιστεύω πως οι Ελβετοί θέλουν να διαρρήξουν τις σχέσεις μας. Αλλά βεβαίω, όπως είπα οι πράξεις έχουν και συνέπειες. Μπορεί να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών αλλά όχι αλλαγή των θεμελιωδών χαρακτηριστικών του και δεν είναι δυνατόν βεβαίως ε, να μιλάνε για μια αμετάκλητη θέση. Ο λαό όμως τη Ελβετία μίλησε, αλλά πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σαφή, Αναμένουμε να διερθούν πλήρω οι συμφωνίε μα. Υπερασπιζόμαστε την αρχή τη ελεύθερη μετακίνηση ω βασική ε, αρχή και αναμένουμε σαφήνεια από του Ελβετού εταίρου μα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Μαγκίνε. Ο κύριος Σβόμποντα για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο ελβετικός λαός μίλησε και πρέπει πράγματι να δεχτούμε την απόφαση αυτή. Αλλά βεβαίως δεν είναι δυνατόν να είμαστε τόσο αφελείς όσο κάποιοι συνάδελφοι και να χαιρόμαστε για το ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλείονται από πιθανές ε, θέσεις εργασίας και δεν είναι δυνατόν βεβαίως να το αποδεχτούμε έτσι απλά. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιους Ελβετούς εδώ πέρα. Αναφέρω από την Neue Zürcher Zeitung, η οποία λέει δεν αποφασίσαμε μόνο μία αλλαγή όσον αφορά τα, το ποιον θα δεχόμαστε στη χώρα, αλλά δεχτήκαμε με το δημοψήφισμα αυτό μία απόφαση αρχής για τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως ας σκεφτούμε ποια ήταν και τα υπόλοιπα δημοψηφίσματα της ε, Ελβετίας. Ε, τελικά θέλουν να έχουν σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε σαφώς στην Ελβετία γιατί εδώ πέρα πρόκειται για ένα πολύ βασικό στοιχείο των ε, σχέσεων μας, όχι κάτι το δευτερεύον το οποίο μπορεί να καταψηφίσουν. Και αυτό είναι και εις βάρος της Ελβετίας, γιατί πάρα πολλοί Ελβετοί εργάζονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα δεχτούμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα τόσο κεντρικό στοιχείο των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας να καταργηθεί. Βεβαίως και στην Ελβετία κάποια στοιχεία οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Π.χ. Ε, υπήρχε και η περίφημη πρωτοβουλία για την καθιέρωση κατώτατου μισθού στην Ελβετία. Δηλαδή υπήρχε οπωσδήποτε και ο κίνδυνος του κοινωνικού ντάμπινγκ στην Ελβετία. Γιατί συχνά υπήρχε ο φόβος ότι θα έρθουν άνθρωποι χωρίς προσόντα οι οποίοι θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των μισθών. Και τέλος, η Ελβετία τελικά φαίνεται ως μια χώρα η οποία θέλει τα λεφτά μας, συχνά και από φοροδιαφυγή, αλλά δεν αποδέχεται τους εργαζόμενους μας. Ε, δεν μπορούμε και εμείς να το δεχτούμε αυτό σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο λεπτά ο κύριος Γκάλαχερ. Ως ναι. πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ελβετία εκ μέρους ε, της ΑΛΤΕ, ε, της πολιτικής ομάδας και εγώ θα πρέπει να εκφράσω την απογοήτευσή μου ε, από τα αποτελέσματα αυτού του πρόσφατου δημοψηφίσματος, βεβαίω θα πρέπει να το αποδεχτούμε, πρόκειται για δημοκρατική απόφαση του ελβετικού λαού. Και η απόφαση που τώρα έχουμε μπροστά μας είναι περίπλοκη, δύσκολη και υπάρχουν πολλές ευαισθησίες και ο συνάδελφος ο οποίος ε, εκράδενε ε, την ελβετική σημαία δεν βοήθησε. Όμως ε, δεν θα πρέπει να κάνουμε κινήσεις εμπριστικές. Είμαστε δεμένοι με αυτή τη χώρα. Πάνω από 60% των εξαγωγών μας πηγαίνουν στην Ελβετία και επίσης έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις η Ελβετία με τη γειτονική Γερμανία και με τις ε, ΗΠΑ και έχουμε μια πρόσφατη μελέτη σε σχέση με το τροπικό σύστημα και λέει ότι 80.000 θέσεις εργασίας ίσως απολεστούν στο μέλλον και η οικονομική ανάπτυξη ίσως ε, φρενάρει ε, στην Ελβετία και κατέβει στο 0,3% άρα θα πρέπει να μην προβούμε σε αντίπεινα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη νέα νομική κατάσταση, θα πρέπει να ενεργήσουμε αναλόγω και θα πρέπει να πούμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Και για τους πρόσφατους από εμάς είναι το θεμελιώδες δικαίωμα τη ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, μια αρχή που ενσωματώνεται στις συνθήκε. Δεν θα πρέπει αυτό να το παραδώσουμε. Η συμμετοχή στο Horizon 2020. Ε, είχαμε μιλήσει και για το Ισραήλ κάποτε. Δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι που να ανατρέψουμε αυτά τα οποία είχαμε αποφασίσει. Οι σχέσεις μας με την ε, χώρα αυτή έχουν πολλές όψεις. Άρα θα πρέπει να προβούμε σε κάποια συμφωνία, μια σφαιρική συμφωνία, κάτι το οποίο το ζητούμε από το 2010 ως Κοινοβούλιο. Είναι κατακλείδη. Απευθύνουμε στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δώσουν διαπραγματευτική εντολή για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος διακόπτει τον ε, κύριο Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Κολμπελίτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Οι Ελβετοί έχουν κάθε ελευθερία να ψηφίσουν όπως θέλουν αλλά είναι υπεύθυνοι και για το αποτέλεσμα της ψήφου τους. Άρα τα πράγματα για μένα είναι απόλυτα σαφή Όλες οι διαπραγματεύσεις με την Ελβετία έχουν διακοπεί και θεωρούμε ότι είναι άκυρες. Δηλαδή βρισκόμαστε στην κατάσταση πριν από τη σύναψη των ε, συμφωνιών. Η Ελβετία θα πρέπει να εξεύρει μια λύση, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελβετική κοινωνία πρέπει να βρει ε, λύσεις γιατί μία εβδομάδα πριν από την ψήφο όλες οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι το 60% θα καταψήφισε εάν είχε κατανοήσει τις συνέπειες. Εμείς πρέπει να αναγνωρίσουμε το αποτέλεσμα της ψήφου. Τους λέμε, είσαστε μεγάλοι, δυνατοί, αυτόνομοι. Ε, βρείτε τα και αν βρείτε μία λύση, ελάτε να μας ξαναβρείτε. θα δείτε ότι οι Ελβετοί θα επανέλθουν γονιπετής, διότι μας χρειάζονται, διότι 60% των εξαγωγών της Ελβετίας μεταβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Αγορά. Δεν μπορούμε να έχουμε τα πάντα και πιστεύω ότι κανένας δεν θα μπορούσε να βρει λύση, ούτε το εθνικό μέτωπο. Είσαστε κρετίνοι, διότι δεν έχετε κατανοήσει τις αξίες της Ευρώπης. Γι' αυτό σας λέω ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να κουνηθεί καν. Έχει συνάψει συμφωνίες, η Ελβετία καταγγέλει τις συμφωνίες, άρα ας βρει η Ελβετία τη λύση και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε χρόνο η Ελβετία θα πρέπει να συντονιστεί με μας. Έτσι έχει η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κονπεντίτ, σας ανακαλώ στην τάξη. Δεν είναι δυνατό να ακούγονται εδώ πέρα λέξεις όπως κρετίνη και ηλίθη. Η Κυρία Φόρντ για μισή λεπτό έχει το λόγο. Η ελευθερία αυτή της μετακίνησης είναι πάρα πολύ σημαντική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ είμαι υπερήφανη όπου ζω στην της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να έρθουν και να μείνουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά πρέπει επίσης να γνωρίσουμε πώς η μετανάστευση μπορεί να ασκήσει πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες και πρέπει να ακούσουμε τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών. Η μετανάστευση ωφελεί την οικονομία μας και όλοι επωφελούμαστε από την γνώση. Πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά και τις δύο πλευρές των επιχειρημάτων. Η Ελβετία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός έχει δικαίωμα να διαλέξει πώς ελέγχει τα σύνορά του. Αλλά πρόκειται για ένα ευαίσθητο ζήτημα και πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι στην απάντησή μας. Η Ελβετία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνεργάζεται μαζί μας σε πολλά ζητήματα. Στην επιστήμη συνεισφέρουν στην χρηματοδότηση της έρευνας και οι ερευνητές τους συμμετέχουν σε συνεργασία στην έρευνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούν να λύσουν προβλήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο και όλοι υποφελούμαστε από την γνώση και την καινοτομία στην οποία συνεισφέρουν και οποιαδήποτε απόπειρα να τιμωρήσουμε την Ελβετία μέσω του περιορισμού της συμμετοχής τους ε, στην ε, έρευνα και την ανάπτυξη θα αποβεί επιζήμια για όλους. Η Ευρώπη αλλάζει. Κάποιες χώρες θέλουν στενότερη ενοποίηση, άλλες όχι. Εάν είναι να μείνουμε όλοι στην ενιαία αγορά, θα πρέπει να επιτρέψουμε σε κάποιες χώρες να μείνουν εκτός κάποιων άλλων κομματιών. Η αντίδραση στο δημοψήφισμα αυτό είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθηθεί πάρα πολύ στενά και θα ήταν νομίζω ανόητο να αντιδράσουμε πάρα πολύ έντονα. Σας ευχαριστώ κύριε Φόρτ. Τον λόγο έχει ο κύριος Τριανταφυλλίδης για ένα λεπτό. Πρόεδρε, στην Ελβετία έχει ληφθεί μια απόφαση που λίγο διαφέρει από τις εξαγγελθήσεις προθέσεις και άλλων χωρών να περιορίσουν την εργασία ξένων στις χώρες τους αυτό συνιστά σαφή διάκριση κατά των μεταναστών εργαζόμενων. οι ξένοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούνται για να μειωθούν τα εργατικά δικαιώματα κυρίω από τι μεγαλοεπιχειρήσεις ω φτηνό εργατικό δυναμικό. τα δικαιώματα του πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστά βάσει των συλλογικών συμβάσεων. Επίση, το βάρο τη κρίση δεν είναι αποδεκτό να φορτώνεται στου εργαζόμενου ντόπιου ή ξένου. αυτό κάνουν σειρά ακροδεξιών έω φασιστικών οργανώσεων και με κάποιο τρόπο και η ευρωπαϊκή ένωση θέτοντας ως προτεραιότητα την ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου σε ολόκληρη την ένωση και μόνο ως δεύτερο ή ως καθόλου προαπαιτούμενο τα δικαιώματα των εργαζομένων. προειδοποιούμε ότι οι δύο αυτές τάσεις αναγεννούν τον φασισμό και τον ρατσισμό. πρέπει να αλλάξει συνολικά η κατεύθυνση σε αυτά τα δύο θέματα τη μετανάστευση και τους εργαζόμενους να καταπολεμηθεί η ασυδοσία των εργοδοτών και η ακροδεξιά ρητορία τα αντίπεινα δεν αποτελούν λύση αλλά χρειάζεται ένα άλλο θεμελιώδης αναπροσανατολισμό για τη μετανάστευση όσο και την προσέγγιση τη εργασία. Στις 9 Φεβρουαρίου 14 ο ελβετικός λαός αποφάσισε για το μέλλον του. Ο ελβετικός λαός ε, είπε να σταματήσει η μετανάστευση. Εμείς λαμβάνουμε γνώση. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε αυτή την ελεύθερη απόφαση. Ε, πιστεύω ότι αν γινόταν το ίδιο δημοψήφισμα σε άλλες χώρες, τι θα γινόταν. Αν ε, γινόταν στην Ιταλία όπου υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια ε, μετανάστες και όπου υπάρχει υψηλός ε, δείκτης ανεργίας και πολλοί Ιταλοί στα στο κατόφλι της φτώχειας, τότε καταλαβαίνετε ότι το δημοψήφισμα θα είχε την ίδια έκβαση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις σωστής επιδοτήσεις που θα πρέπει να δοθούν προς τους Ιταλούς. Δεν μπορούμε να, δεν μπορούν να ζητάνε οι μετανάστες τα πάντα χωρίς ε, να προσφέρουν τίποτα. 5 εκατομμύρια Ιταλοί δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας διότι δεν έχουν χρήματα. Νομίζω ότι οι δικοί μας πολίτες δεν δέχονται την υπεροψία αυτής της Ευρώπης που θέλει να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της Ευρώπης. Τη στιγμή που δεν υπάρχει εργασία για τους δικούς μας πολίτες και τη στιγμή που δεν διασφαλίζουμε υπηρεσίες για τους ε, δικούς μας πολίτες, οι μετανάστες θα πρέπει να παραμείνουν εκτός. Δεν πρόκειται για ρατσισμό. Είναι ο λάθος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Η Ευρώπη δείχνει την ανικανότητά της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ, Κλέρις, για ένα λεπτό. Τι θλιβερό θέαμα ήταν αυτή η συζήτηση. Έπρεπε να το δείχνουμε στην τηλεόραση για να τα ακούν αυτά οι ψηφοφόροι. Να βλέπουν τον αυταρχικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αποξενωθεί από τους λαούς. Συζητάμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε το αποτέλεσμα ενός δημοκρατικού δημοψήφισματος. Όχι, κύριε Κονμπεντίτ. Δεν είναι αυτό το οποίο νομίζετε. Το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος για τη μαζική μετανάστευση είναι το ότι ένας λαός θέλει να είναι το αφεντικό στη χώρα του και να αποφασίζει ποιος θα μπαίνει. Δεν έχει ουδεμία σχέση με ξενοφοβία. Είναι λογική αντίληψη και εύχομαι να έχουμε τέτοια δημοψίσματα στη Φλάνδρα, στην Ολλανδία, στη Γαλλία και αν γίνουν θα έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά μην ανησυχείτε, έρχεται η 25η Μαΐου. Σας ευχαριστώ. Εδώ τελείωσε ο κατάλογος των ομιλητών. Τώρα για την Κομισιόν ο κύριος Επίτροπος. Ε, ε. κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ. Όπω μια σειρά βουλευτών ε, προανέφεραν, η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και το δικαίωμα παροχή υπηρεσιών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία ισχύουν πολύ χρόνο από το 2002. Οπότε αυτό έχει δημιουργήσει και για τις δύο πλευρές ωφέλεια, οπότε ε, Βεβαίω, η Ελβετία είναι στο κέντρο τη Ευρώπη ε, έχουμε τι ίδιε κοινέ αξίε, έχουμε τι ίδιε προκλήσει να αντιμετωπίσουμε, οπότε το μέλλον της Ελβετία ε, είναι στην Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει η Ελβετία να αντιδράσει σε σχέση με το δημοψήφισμα. Αλλά θα πρέπει να εργαστούμε χέρι-χέρι με την Ελβετική κυβέρνηση και θα πρέπει σε καινούργια βάση να οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας στο μέλλον να είναι προς όφελος και των δύο πλευρών. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για το Συμβούλιο, κύριε Σκουρκούλας. Thank you, President. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, όπως μόλις είπε η Κομισιόν, έχουμε παραδοσιακές και ισχυρές σχέσεις με την Ελβετία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος, οι οικονομίες μας είναι στενά συνδεδεμένες, αλλά πρέπει να επαναλάβουμε πως η ελεύθερη μετακίνηση είναι μία από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες, είναι θεμελίος λίθος εσωτερικής αγοράς και πρέπει να είναι σαφές πως δεν μπορούμε να διαλέγουμε ποια από αυτές τις ελευθερίες μας αρέσει. Είναι πακέτο και πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη-μέλη και τους εταίρους. Σεβόμαστε πλήρω. την απόφαση του ελβετικού λαού, αλλά βεβαίως αναμένουμε και από την Ελβετία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις συμφωνίες. Να αναφερθώ σε ένα σημαντικό ζήτημα. Το Συμβούλιο παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα όσα αναφέρονται στον τύπο και τις ε, πρόσφατες επιθέσεις στην ελευθερία της μετακίνησης. Θεωρούμε πως οι γενικεύσεις και αυτά τα οποία αναφέρονται για πατεώνες και για αυτούς οι οποίοι κάνουν τουρισμό επιδομάτων είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, ειδικά υπό το φως του λαϊκισμού. Ως πολιτικοί πρέπει να μην ενδώσουμε στις λαϊκιστικές και ξενοφοβικές τάσεις. Η αντίληψη κοινή γνώμη σχετίζεται άμεσα με τι πολιτικέ δηλώσει και πρέπει οι κατηγορίε να βασίζονται σε στοιχεία και νούμερα και όχι σε κάποιε αντιλήψει. Σα ευχαριστούμε κύριε Κούρκουλα. Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλο τη συζήτηση για αυτό το θέμα τη ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Γκόλνη θέλει τον λόγο για μια προσωπική παρατήρηση. Έχετε, κύριε Γκολνή. σας Υπενθυμίζω όμως πως σύμφωνα με τον κανονισμό